Παρακαλώ καθίστε. Γιατί δεν μπορούμε να κρατήσουμε την για πολλή ώρα. Έπονται άλλοι. Παρακαλώ καθίστε λοιπόν. Καλημέρα. Καλημέρα σε όλες και όλους. Καλημέρα στα μέλη της Επιτροπής μας ε, και τα παλαιότερα, κάποια που βλέπω τουλάχιστον, και στα νέα να ευχηθώ. Καλώς ήρθατε. Έχουμε και τις εκπροσώπους της Επιτροπής ε, που θα μας συνοδεύουν σε όλη αυτή την κοινοβουλευτική περίοδο. Φαντάζομαι υπάρχουν εδώ εκπρόσωποι και της Κομισιόν του Συμβουλίου. Βέβαια και τη γραμματεία να την καλωσορίσω και τους συνεργάτες μας. Να σας καθησυχάσω ότι δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ε, από την αρχή την Διατλαντική Συμφωνία. Λοιπόν, είναι σύντομη όπως βλέπετε η μερική διάταξη και ελπίζω οι εργασίες να κυλήσουν ομαλά. Το βασικό θέμα της μερικής διάταξης φυσικά είναι η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής. Και θα ξεκινήσουμε με την εκλογή του Προέδρου της Επιτροπής μας. Κυρίσω λοιπόν την έναρξη της ε, συνεδρίασης συγκρότησης σε σώμα. Θέλω να επιθυμίσω στους βουλευτές ότι θα εκλέξουμε τον Πρόεδρο και τους Αντιπροέδρους της Επιτροπής αυτής. Πρώτα τον Πρόεδρο και μετά τους Αντιπροέδρους. Ο κύριος Ντάρτμουθ, γνωστός στους παλαιότερους. Ε, κύριε Ντάρτμουθ, θέλετε το λόγο για τον κανονισμό, έχετε έτοιμο από τη Για ποιο άρθρο παρακαλώ. Um, I would Πριν την εκλογή του νέου Προέδρου και των νέων Αντιπροέδρων, θα ήθελα να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή Μορέιρα, τον ε, περχόμενο πρόεδρο, απελθόντα πρόεδρο, ο οποίος νομίζω ότι με πάρα πολύ μεγάλο επαγγελματισμό γύθηκε των εργασιών της Επιτροπής μας και νομίζω ότι θα έπρεπε να τον ευχαριστήσουμε. Ήθελα να το βάλω και στην σχεδιάταξη, αλλά δεν υπήρχε χρόνος. Θα στείλουμε, λέει ο πρόεδρος, ένα μήνυμα εξ όλων των μελών θα στείλουμε λοιπόν τις ευχαριστίες μας και τα συγχαρητήριά μας στον πρόεδρο Μορέιρα. Και τώρα να σας ανακοινώσω τον κατάλογο των αναπληρωματικών μελών που αντικαθιστούν τακτικά μέλη που δεν είναι σήμερα παρόντα. Ο κύριος Βαλέσα αντικαθιστά τον κύριο Κασπάρη, ο κύριος Μάτο τον κύριο Φέλνερ, ο κύριος Σάτσερ ή Ζάχερ τον κύριο Λαντσμπέργκης, ο κύριο Βαντενκάμπ, τον κύριο Πάπριτς, ο κύριος Κέλλη, την κυρία Κβίστοντ Ρόβολ, ο Ερίκ Αντριέ, τον κύριο Λίνκφρετ. για του ECR, κύριο Σταρμπάτη, αντικαθιστά τον κύριο Κάμπελ Μπένερμαν, για την Άλντε. Η κυρία Σαρών Σοβά αντικαθιστά την Μαριάν Ντε Σαρνές και ο κύριος Βαν τον κύριο Λάνσδορφ. Για τους μη γεγραμμένους. κύριο Σόχρατ, την κυρία Λεπέν. Α, είστε εδώ κύριε Λεπέν. Δεν έχουμε το σωστό κατάλογο, από ό,τι φαίνεται. Ο κύριος Επιτίδιος θα τον κύριο Μπερμάιε και ο κύριος Ντεγκράφ, τον κύριο Σαλπίνη. Ολοκληρώνω λοιπόν. Αυτές είναι οι... Αυτοί είναι οι αντικαταστάτες και είναι σημαντικό να το ξέρουμε σε περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάποια ψηφοφορία. Να υπενθυμίσω σε όλους σας ότι θα πρέπει να έχετε μαζί σας την κάρτα ψηφοφορίας αν όχι φαντάζομαι ότι ήρθε σε επαφή μαζί σας ε, κάποιος από τη γραμματεία και αν δεν έχετε την κάρτα σας πρέπει να ρυθμιστεί αυτό το θέμα. Έχετε καταρχάς όλοι μαζί τις κάρτες. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε λοιπόν στην εκλογή του Προέδρου ή της Προέδρου της Επιτροπής αυτής. Έχουμε απαρτία. Είναι εδώ 11 μέλη, πάνω από το 1 τέταρτο δηλαδή. Το ξεπερνάμε κατά πολύ. Υποψηφιότητες λοιπόν για τη θέση του ή της Προέδρου της Επιτροπής μας παρακαλώ. Να δώσω το λόγο στον ε, David Μάρτιν από την ε, Σοσιαλιστική Ομάδα. Σε ευχαριστώ Γιάννικ και σε ευχαριστώ που ασκείς πολύ επιτυχημένα την Προεδρία μέχρι τώρα. Δεν θα κρατήσει πολύ, λέει ο κύριος Ζαντό. Ε, γι' αυτό το λέω, λέει ο κύριος Μάρτιν. Τον Μπέρτ Λάγκε θα ήθελα να προτείνω Όσοι ήταν ήδη εδώ γνωρίζουν ότι έχει εμπειρία για να προεδρεύσει τη Επιτροπή σαν συντονιστή τα τελευταία πέντε χρόνια για τη Σοσιαλιστική Ομάδα. Είναι μέλο του Κοινοβουλίου 15 χρόνια, είναι ευφυή, ε, έχει κίνητρα, έχει ίσω και σημαντικότερο υπομονή και χιούμορ για την Επιτροπή μα και τι πολύ ενδιαφέρουσε συζητήσει. Λοιπόν, πρότασή μα Μπέρντ Λάγκε. Πρόεδρος, περίμενα κάποιες κριτικές να ακούσω τίποτα, όλα θετικά. Ε, για τον υποψήφιο. Ωραία. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, παρακαλώ, άλλες προτάσεις. Όχι. Επομένως, σας προτείνω. Πρώτα απ' όλα να ρωτήσω αν έχετε κάνει τη δήλωση χρηματοοικονομικών συμφερόντων, κύριε Λάγκε. Δέχεστε την υποψηφιότητα, συμφωνείτε με την υποψηφιότητά σα εκ μέρου ομάδα και του κ. Μάρτιν, συμφωνείτε. Είστε μέλο τη Επιτροπή. Τακτικό, ναι. Άρα σα προτείνω, αγαπητοί συνάδελφοι, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, να εγκρίνουμε διαβοή την υποψηφιότητα. Τον ορισμό του κ. Λάγκη δηλαδή. Στη θέση του Πρόεδρου, Μπέντ Λάγκε, έλα να καθίσει στη θέση μου, στην παραχωρώ. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Ganz herzlichen Dank für das entgegengebrachte. Συνάδελφοι, σας ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη σας. Υπόσχομαι να κάνω ό,τι περνά από το χέρι μου ώστε να σας αποδείξω ότι σωστά μου δώσατε την εμπιστοσύνη σας και δικαίως. Στην Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου Έχουμε πολλές ευθύνες και θα είμαστε πολύ απασχολημένοι στην επόμενη πενταετία. Έχουμε να ασχοληθούμε με την επερχόμενη συμφωνία και ελπίζω πως επί τη βάση ενός επικοδομητικού διαλόγου θα μπορέσουμε να σημειώσουμε πρόεδρο, ε, πρόοδο. Λοιπόν, πρώτο μας ε, καθήκον είναι να πληρώσουμε τα θέσει του Προεδρείου. Οπότε θα προχωρήσουμε στην εκλογή του πρώτου Αντιπροέδρου της Επιτροπής. Έχουμε εξετάσει τον κατάλογο των μελών. Έχουμε απαρτία. 11 είναι το μήνυμο μελών που πρέπει να είναι παρόντα και γι' αυτό θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχουν υποψηφιότητες για την πρώτη αντιπροεδρία αυτής της Επιτροπής. Κύριε Βίνκλερ, σας ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και πριν να παρουσιάσω τον υποψήφιο, θέλω να σας συγχαρώ που αναλάβατε την Προεδρία αυτής της Επιτροπής εξ ονόματος της ομάδας του ΕΛΚΑ. Έχω την χαρά και την τιμή τώρα να προτείνω την υποψηφιότητα της κυρίας Τόκια Σαΐφη ως πρώτης Αντιπροέδρου της Επιτροπής ΙΝΤΑ. Η συνάδελφος Τόκια Σαΐφη είναι γνωστή στα μέλη της Επιτροπής Ίντα, είναι μέλος αυτής της Επιτροπής από τότε που συστάθηκε το 2004. Επίσης ε, διετέλεσε ε, τη συντονίστρια της ομάδας του ΕΛΚ τα τελευταία θητεία και έχει υπάρξει συγγήτρια ή σκιώδηση συγγήτρια για πολλούς σημαντικούς φακέλους στην τελευταία εντολή και επίσης διατέλεσε πρόεδρος της Επιτροπής της Πολιτικής Επιτροπής της Συνέλευσης ΕΡΟΜΕΔ πριν να έρθει δε στο Ευρωκοινοβούλιο ήταν υφυπουργό για τη βιώσιμη ανάπτυξη στο πλαίσιο της γαλλικής κυβέρνησης. Θα ολοκληρώσω λέγοντας ότι είμαι βέβαιος ότι θα παίξει σημαντικό ρόλο στο Προεδρείο της Επιτροπής μας και θα βοηθήσει στην αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα των εργασιών μας. Ευχαριστώ. Θα ευχαριστώ πολύ για την πρόταση αυτή. Υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Ε, όχι. Οπότε θα στραφώ στην κυρία Σαΐφη τώρα. Έχετε συμπληρώσει την δήλωση χρηματοοικονομικών συμφερόντων σας, να έχετε υποβάλει και έπειτα να ρωτήσω και αν είστε τακτικό μέλος της Επιτροπής, επίσης εάν δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, ναι και στις τρεις ερωτήσεις. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Σαΐφη. Τώρα... Να ρωτήσω. Αν διαβοής μπορούμε να εκλέξουμε την πρώτη αντιπρόεδρο. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Dann herzlichen Glückwunsch, Frau Sifi, auf gute Zusammenarbeit und bitte Kommen Συγχαρητήρια κυρία Σαΐφη, παρακαλώ ελάτε εδώ στα έδρανα του Προεδρείου. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann kommen wir Ωραία, λοιπόν, συνάδελφοι, προχωρούμε τώρα στην εκλογή του δεύτερου αντιπροέδρου της Επιτροπής. Υποψήφιοι, κυρία Κέλλορ, σας ευχαριστώ, συγχαρητήρια και στους δύο σας για την εκλογή σας. Θα ήθελα να προτείνω εξ ονόματος των Πρασίνων τον Γιάννικ Ζαντό για τη δεύτερη αντιπροεδρία αυτής της Επιτροπής. Όλοι γνωρίζετε τον Νίκη Ζαντό ότι είναι πολύ αφοσιωμένο μέλος αυτής της Επιτροπής και εργάζεται εδώ και πολλά χρόνια για εμπορικά θέματα από το 1994 όπου εργάστηκε και εντός της Greenpeace πολύ γνώστης του, του θέματος λοιπόν και θα ήμουν ευτυχής αν μπορούσατε να τον υποστηρίξετε ως δεύτερο αντιπρόεδρο της ΙΝΤΑ. Ευχαριστώ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Άλλες υποψηφιότητες υπάρχουν. Από ό,τι φαίνεται όχι. Τις τρεις ίδιες ερωτήσεις έχω να σας υποβάλω, Γιάννη. Έχετε υποβάλει τη ε, δήλωση συμφερόντων, είστε πλήρε, ε, τακτικό μέλος και ε, δέχεστε την υποψηφιότητα αυτή. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Και για τις τρεις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ζαντό. Τέλος, διαβοής μπορούμε να εκλέξουμε τον δεύτερο αντιπρόεδρο. Σας ευχαριστώ πολύ και συγχαρητήρια νικ Μπορείς να έρθεις στο Προεδρείο. das Präsidium zu vervollständigen, geht es um die Wahl des oder Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε στην εκλογή του τρίτου αντιπροέδρου. Έχουμε, εξακολουθούμε να έχουμε απαρτία. Υποψηφιότητες. Παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν να σας συγχαρώ για την εκλογή σας και να συγχωρώ τον Γιάννη Κιζαντό για την Αντιπροεδρία. Θα ήθελα εξ ονόματος του ΕΛΚ να σας πω πως έχω την τιμή και τη χαρά να σας υποβάλω την υποψηφιότητα του Χούλιο Βίνκλερ για την θέση του τρίτου Αντιπροέδρου. Ο κύριος Βίνκλερ είναι μέλος της Επιτροπής ΙΝΤΑ από το 2007. Ε, είναι αναγνωρισμένος από πολλούς συναδέλφους αυτής της Επιτροπής για το εξωσημείο του έργο του και για την ε, παρακολούθηση των υποθέσεων που αφορούν τα Δυτικά Βαλκάνια. Πριν να έρθει στο Ευρωκοινοβούλιο, ο κύριος Βίνκλερ διατέλεσε Υπουργό Εμπορίου της Ρουμανίας από το 2004 μέχρι το 2007 και Υπουργό Επικοινωνίας και Τεχνολογίας κατά τη διάρκεια του 2007. Είμαι βεβαία ότι η παρουσία του κυρίου Βίνκλερ στην ομάδα θα είναι πλεονέκτημα για τις εργασίες μας. Σας ευχαριστώ. Ganz Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή την πρόταση. Υπάρχει άλλη υποψηφιότητα. Όχι. Κύριε Βίνκλερ, τρεις ερωτήσεις. Έχετε υποβάλει την δήλωση συμφερόντων, είστε τακτικό μέλος και δέχεστε την υποψηφιότητα. Μάλιστα, Πρόεδρε. Είμαι μέλος, έχω υπο... Ε, τακτικό μέλος, ε, έχω υποβάλει τη δήλωσή μου και θα είναι τιμή μου να είμαι μέλος του Προεδρείου και να συνεργαστώ μαζί σας. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ. Μπορούμε διαβοής να εκλέξουμε τον τρίτο αντιπρόεδρο. Ganz herzlichen Glückwunsch, Herr Winkler. Σας ευχαριστώ πολύ. Συγχαρητήρια κύριε Winkler. Θα ήθελα να σας ζητήσω τώρα να έρθετε κι εσείς εδώ στο Προεδρείο. Και έτσι είναι πλήρως το Προεδρείο μας. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das Präsidium ist vollständig und ich bin mir sicher, dass wir gemeinsam Κυρίες και κύριοι, είναι πλήρες τώρα το Προεδρείο μας. Α, με συγχωρείτε. Έχουμε να εκλέξουμε και τον τέταρτο αντιπρόεδρο, τον Ιτίν, τέταρτο αντιπρόεδρο. Η ίδια διαδικασία θα ακολουθήσουμε, την ίδια μάλλον διαδικασία. Έχουμε απαρτία, έχουμε καταγράψει τα αναπληρωματικά μέλη, έχουμε υποψήφιο, υποψηφίους για τη θέση του τέταρτου αντιπρόεδρου. Μάλιστα, Έμα, Ευχαριστώ Πρόεδρε και συγχαρητήρια σε εσά και στου αντιπροεδρου. Και εγώ ανησυχούσα ότι ξεχάσαμε τον τέταρτο αντιπρόεδρο, αλλά βλέπω πως έχει κενωθεί μια θέση εκεί στο Προεδρείο. Γι' αυτό θέλω να προτείνω τον συνάδελφο Γιάν Ζαρεντό από την Τσεχία. Είναι μέλος της Επιτροπής τα τελευταία πέντε χρόνια και νομίζω θα είναι εξαιρετική προσθήκη στο Προεδρείο. Ελπίζω πως και εσείς θα βοηθήσετε ε, στην υποψηφιότητα του Γιάννη Ζαραντήλ από το ECR. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρότασή σας. Λέγαμε νωρίτερα ότι θα συνεργαζόμασταν πολύ καλά μαζί. Τις τρεις ίδιες ερωτήσεις έχω να υποβάλω. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλος υποψήφιος. Έχετε υποβάλει την δήλωση συμφερόντος σας, είστε τακτικό μέλος και δέχεστε την υποψηφιότητα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ναι, έχω όντως ε, κάνει την δήλωση συμφερόντων. Είμαι πλήρε, ε, τακτικό μέλος της Επιτροπής και είναι τιμή μου να είμαι στο Προεδρείο μαζί σας. Δέχομαι λοιπόν την υποψηφιότητα. Και σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Ζάχρεντιλ, για μπορούμε να εκλέξουμε τον τέταρτο αντιπρόεδρο. Ja, Σας ευχαριστούμε πολύ, αγαπητοί συνάδελφοι. Τώρα μπορούμε να πούμε ότι είναι πλήρε πλέον το Προεδρείο. Οπότε μπορούμε πλέον να αναλάβουμε δράση και να κατευθύνουμε το σκάφος στο οποίο όλοι βρισκόμαστε μέσα από την καταιγίδα που ενδεχομένως θα έρθει ή δεν θα έρθει. Για τις ημερομηνίε τώρα, για το χρονοδιάγραμμα των συνεδριάσεων, μέχρι το τέλος ε, του έτους έχετε ένα κατάλογο, αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θεωρούμε ότι εγκρίνεται το χρονοδιάγραμμα. Και να σας επισημάνω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας ε, είναι στις 3 το μεσημέρι στις 22 Ιουλίου. Θα πρέπει να λάβουμε και κάποιες αποφάσεις ε, αρχής, αλλά θα έρθει και ο αρμόδιος επίτροπος, στον οποίο θα θέσουμε ερωτήσεις και συγκεκριμένα ο κύριος Ντεχούχτ. Έχετε λοιπόν τον κατάλογο, τον πλήρ θα τον λάβετε όλοι. Αναπληρωτές και τακτικά μέλη. Τέταρτο σημείο, γλωσσικό προφίλ. Επειδή δεν έχουν οριστεί όλοι οι αναπληρωτές, δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα σήμερα. Θα πρέπει να το αναβάλουμε για τις 22 Ιουλίου. Τότε θα λάβουμε την απόφαση για το γλωσσικό καθεστώς. Θα έχουμε τότε όλους τους αναπληρωτές. Σας παρακαλώ λοιπόν και στρέφομαι σε όλες τις πολιτικές ομάδες να ορίσετε τάχιστα τα αναπληρωματικά μέλη. Σημείο 5. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Δεν έχω σήμερα ανακοινώσεις. Το μόνο που θέλω να πω πολύ ξεκάθαρα είναι ότι θέλω ε, να προεδρεύσω σε συνεργασία με όλους σας. Αυτό είναι το πνεύμα που θα με διέπει ως πρόεδρο. Εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το γνωρίζουν οι παλαιότεροι, Ενίοτε διαφωνούμε με άλλες επιτροπές για το ποια κατεύθυνση πρέπει να ακολουθήσουμε, μπορεί να υπάρχει σύγκρουση αρμοδιοτήτων. Εμείς, δυνάμει της συνδική της Λισαβόνας, έχουμε ως Επιτροπή πολλές αρμοδιότητες και νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε πολύ θετικά στην περαιτέρω εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πλέον μια μεγάλη Επιτροπή, 41 μέλη. Σίγουρα θα απαιτηθεί πολλή δουλειά από όλους μας, πολλά έχουμε να κάνουμε, ιδίως σε θέματα πνευματικής ιδιοκτησίας ε, εντός Ευρώπης αλλά και ε, όχι μόνο. Ελπίζω να μπορέσουμε να προασπίσουμε αποτελεσματικά τα ευρωπαϊκά συμφέροντα. Πρέπει να σας πω ότι πολλές εμπορικές συμφωνίες ε, τα τελευταία δύο χρόνια συζητήθηκαν ίσως και κλεισμένο των θυρών σε πολλές περιπτώσεις γιατί δεν Υπήρχε πολύ ενδιαφέρον. Τώρα όμως έχουν αλλάξει τα πράγματα. Υπάρχει και πολύ μεγαλύτερο ενδιαφέρον και μεγαλύτερος έλεγχος. Η εμπορική πολιτική είναι πολύ σημαντική. Είναι ένα σημαντικό τομέα ε, για την Ευρωπαϊκή Ένωση και όχι μόνο. Και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης το εμπόριο έχει πολύ μεγάλη σημασία, άρα πρέπει να είναι στο επίκεντρο των πολιτικών συζητήσεων. επομένω και η κοινωνία των πολιτών αλλά και τα πολιτικά κόμματα θα πρέπει να συμμετέχουν στη συζήτηση και στις διαβουλεύσεις για τις διάφορες εμπορικές συμφωνίες, TTIP, TISA. Πρέπει και εμείς να έχουμε λόγο, να αρθρώσουμε και για μένα είναι μια ε, ευκαιρία να δώσω μεγαλύτερη διαφάνεια σε όλες αυτές τις συζητήσεις. ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες και να μην θεωρηθεί ε, κανείς ότι μένει εκτός. Δεν θέλουμε να είναι μόνο ελεύθερη η εμπορική πολιτική, αλλά και δίκαιη. Και αυτό είναι ένα σημαντικό σημείο προσυζήτηση. Πώς μπορούμε να το πετύχουμε, γιατί θέλουμε να δούμε τις ίδιες τις συμφωνίες και το περιεχόμενό τους, αλλά και την ίδια την ουσία της δίκαιης εμπορικής πολιτικής. Αυτά προς το παρόν δεν θέλω να επεκταθώ περισσότερο σήμερα τουλάχιστον. Θα έχουμε, ελπίζω, επικοδομητική συνεργασία. Αυτός είναι ο δικός μου στόχος. Παρακαλώ, ποιος θέλει το λόγο για δικαστικό. Ο κύριος Ντάρθμουθ. Ναι, πολύ σωστά μιλήσατε για τη μεγάλη δουλειά που περιμένει την Επιτροπή μας και τις πολλές αρμοδιότητες που έχουμε δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Αυτό το πλαίσιο, στο χρονοδιάγραμμα ε, βλέπω έτσι ελαφρύ κάπως το πρόγραμμα. Έχουμε τη συμφωνία TTIP, έχουμε πολλά άλλα να συζητήσουμε. Δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη, ε, το κατάλληλο μέρος για να προτείνουμε μια αναδιάρθρωση, μια αναδιοργάνωση του χρονοδιαγράμματος. Απλά θέλω να το σκεφτείτε αυτό, λαμβάνοντας υπόψη τις αρμοδιότητές μας και τα διάφορα άλλα στις διάφορες υποχρεώσεις που έχουμε. Ο πρόεδρος, ναι, πράγματι θα τα δούμε, θα τα συστήσουμε και στην επόμενη συνέντευξη των συντονιστών μας στις 22 Ιουλίου όλα αυτά τα θέματα. Και αν δεν αρκούν θα πρέπει να συμφωνήσουμε για παραπάνω συνεδριάσεις. Προς το παρόν αυτά λοιπόν, κάθε επιτυχία σε όλους, καλή ημέρα, καλό υπόλοιπο.